Cari colleghi, αγαπητοί συνάδελφοι, με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση θα μου επιτρέψετε να καλωσορίζω στην σημερινή μας Ολομέλεια τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω για την επίσκεψή σας εδώ. Είναι μεγάλη τιμή για μας το ότι επιλέξατε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη δεύτερη έξοδό σας από την Γερμανία στα πλαίσια του νέου σας ρόλου μετά από αυτήν στο Παρίσι την προηγούμενη εβδομάδα και μόνο ούτε τρεις εβδομάδες από την ημέρα που αναλάβατε τη νέα σας θέση. Η παρουσία σας εδώ λοιπόν δείχνει την αφοσίωσή σας στην Ευρώπη, την ισχυρή αφοσίωσή σας. Ζητήσατε περισσότερο θάρρος για την Ευρώπη, για μια καλύτερη Ευρώπη, ελεύθερη Ευρώπη, Ευρώπη εργασίας, ευημερίας και δικαιοσύνης. Είμαι λοιπόν πεπισμένος ότι το θάρρος το οποίο αναζητείτε μπορείτε να το βρείτε ανάμεσα στα μέλη αυτού εδώ του Κοινοβουλίου. Με την παρουσία σας λοιπόν κύριε Πρόεδρε υπενθυμίζετε και την αφοσίωση της χώρας σας για την Ευρώπη, μια πολύ σημαντική προσπάθεια ιδιαίτερα μετά από την απόφαση ενός κράτους μέλους να εξέλθει της Ενώσεως. Βιώνουμε δύσκολες στιγμές, έχουμε ζήσει αντίστοιχες στιγμές και στο παρελθόν και πάντα η πολιτική μας ένωση βρήκε την κατάλληλη λύση με τα κατάλληλα μέτρα. Αγαπητέ Πρόεδρε, δεν θα σας ζητήσω να δώσετε λεπτομερείς απαντήσεις σήμερα, αλλά θα σας ζητήσω να εργαστείτε μαζί μας για το κοινό μας μέλλον. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για την παρουσία σας κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Αντώνιο, αγαπητοί βουλευτές, ε, κύριε Πρόεδρε της Κομισιόν, αγαπητέ Ζαν Κλοντ, κυρίες και κύριοι. Είναι πραγματικά χαρά και τιμή μου σήμερα που βρίσκομαι εδώ σε αυτόν τον τόπο του ελεύθερου λόγου και του ανοιχτού διαλόγου. Αλλά, αγαπητοί μου φίλοι, η χαρά μου βεβαίως σκιάζεται γιατί υπάρχει πραγματικά πικρία για το ότι μιλάω σε αυτή την Ολομέλεια για πρώτη φορά μετά την αποχώρηση ενός κράτους μέλους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πραγματικά πικρό και με πικραίνει όχι μόνο ως πολιτικό αλλά πρώτα απ' όλα ως πολίτη της Ευρώπης. Εγώ έχω περίπου την ηλικία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν γεννήθηκα το 1956 σε ολόκληρη την Ευρώπη οι πόλεις μας ακόμα είχαν τις πληγές του πολέμου που ξεκίνησε η Χιτλερική Γερμανία. Και ακόμα μεγαλύτερες ήταν οι πληγές στις καρδιές των γειτόνων μας. Και όμως τότε έδωσαν το χέρι τότε στην χώρα μου για να προχωρήσουμε εν ειρήνη στη Ρώμη πριν από 60 χρόνια και έτσι έθεσαν τα θεμέλια για τη Νέα Ευρώπη. Όταν πήγα στο σχολείο, ήδη οι νέοι πριόνιζαν συμβολικά τις μπάρε στα ευρωπαϊκά σύνορα για να πούν θέλουμε περισσότερη Ευρώπη. Και δεν μας αρκεί αυτό το οποίο κάνετε. Το 1968 καταργήθηκαν τα τελωνία εντός της Ευρώπης και σταμάτησαν οι τεράστιες ουρές των φορτηγών στα σύνορα και έγιναν πιο μικρές οι ουρές των γιοταχή. Όταν πήγα στο πανεπιστήμιο η έλξη της Ευρώπης ήταν τόσο μεγάλη ώστε οι άνθρωποι στον νότο της Ευρώπης, στην Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ισπανία δεν έριξαν μόνο τις δικτατορίες αλλά ακολούθησαν μια πορεία ελευθερίας και δημοκρατίας εντός της Ευρώπης. Το 1989 ήμουν στην τελευταία φάση του διδακτορικού μου όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου, το οποίο έριξαν οι θαραλέοι άνθρωποι της Ανατολικής Ευρώπης με ειρηνικό τρόπο για να κατακτήσουμε την ελευθερία και την δημοκρατία. Αυτοί ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι εξασφάνισαν όχι μόνο την ενότητα της χώρας μου, αλλά την επανενοποίηση της Ευρώπης. Κυρίε και κύριοι, όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εννοούμε όταν λέμε στην διακήρυξη της Ρώμης ότι η τύχη μας είναι κοινή. Όλα αυτά είναι η μεγάλη κληρονομιά που μας κληροδότησαν οι μητέρες και οι πατέρες της Ευρώπης. Η πολύτιμη αυτή κληρονομιά, την οποία δεν μπορούμε να αφήσουμε στους εχθρούς της Ευρώπης. Πρέπει να την διατηρήσουμε, να την βελτιώσουμε αυτή είναι η κοινή ιστορική μας αποστολή. Κοιτώντας τα 60 χρόνια της ζωής μου και την ίδια χρονική περίοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε βλέπουμε ακριβώς πώς μεγάλωσε και δημιουργήθηκε η νέα Ευρώπη. Ο δρόμος που διασχίσαμε από τα δελτία της μεταπολεμικής Ευρώπης μέχρι το να γίνει η Ευρώπη η ελπίδα για έναν πιο δίκαιο και ειρηνικό κόσμο. Σε κάποιους μοιάζει σαν τα επιτεύγματα αυτά να είναι μόνιμα και εγγυημένα. Αλλά στη ζωή μου εγώ είδα και τα προβλήματα της Ευρώπης, τις κρίσεις, τις αντιφάσεις, τις οπισθοχωρήσεις και θεωρώ και σε αυτό συμφωνούν και πολλοί άνθρωποι της γενιάς μου πως ο δρόμος της Ευρώπης, της ευρωπαϊκής ενοποίησης δεν μπορεί να πάει προς τα πίσω. Αυτό όμως ήταν ένα λάθος. Όχι. Το μέλλον της Ευρώπης δεν είναι βέβαιο. Ποτέ δεν ήταν βέβαιο. Και δεν χρειαζόταν τον Brexit για να το διαπιστώσουμε αυτό. Θυμάμαι, κυρίε και κύριοι, το 2005. Ήμουν υπουργό εσωτερικών της χώρας μου και εκεί πέρα τότε απέτυχε το όνειρο του Ευρωπαϊκού Συντάγματος. Και ξέρω πάρα πολύ καλά πόσο απογοητευμένοι ήταν πολλοί από εμάς και γνωρίζω εξίσου καλά πως εμείς και πολλοί από εσάς υποθέτω σε αυτή την αίθουσα προσπαθήσαμε και κάναμε αυτό το οποίο κάνει πολύ καλά η Ευρώπη. Συνεχίσαμε. Πήραμε τα τηλέφωνα, ακούσαμε ο ένας τον άλλον, καθίσαμε όλη νύχτα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και κομμάτι-κομμάτι φτιάξαμε τη συνθήκη της Λισαβόνας. Τι θέλω να πω, κυρίε και κύριοι. Η Ευρώπη δεν ήταν ποτέ περίπατος. Η Ευρώπη είναι ένα περίπλοκο και δύσκολο έργο, αλλά αξίζει ο κόπος. Δεν πρέπει να μας πείσουν αυτοί οι οποίοι βρίζουν την Ευρώπη. Η συνεργασία, η αυξανόμενη ευημερία και κυρίως τα 70 χρόνια ειρήνης. Αυτή είναι η υπόσχεση της Ευρώπης. Αλλά βεβαίω αυτή η υπόσχεση δεν εκπληρώθηκε ποτέ από μόνη της. Εκπληρώθηκε όταν ξεπεράσαμε την εθνική στενομυαλιά και φτάσαμε στην ευρωπαϊκή λογική. Και γι' αυτό ακριβώς ήρθα σήμερα σε σας. Ήθελα ο πρώτος μου λόγος ως πρόεδρος της Γερμανίας εκτός της χώρας να γίνει εδώ, σε αυτό το κοινοβούλιο. Ειδικά τώρα, σε καιρούς αυξανόμενων φυγόκεντρων δυνάμεων, από, που έχουμε προφήτες της καταστροφής θα ήθελα εγώ να πάρω το, μέτρο, το μέρος της Ευρώπης. Ως πολίτες, όπως και πολλοί πολίτες τις τελευταίες εβδομάδες, έτσι και εγώ πρέπει να πω ότι ναι θέλω την Ευρώπη, ναι η μεγάλη πλειοψηφία των Γερμανών θέλει την Ευρώπη. Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στο άσχημο παρελθόν. Θέλουμε τον κοινό δρόμο προς ένα καλύτερο ευρωπαϊκό μέλλον. Και όταν λέμε ναι στην Ευρώπη, δεν πρέπει βεβαίως να λέμε ότι τα πράγματα είναι ρόδινα. Όποιος λέει ναι στην Ευρώπη, λέει ναι και στα περίπλοκα, στα κουραστικά και στα δύσκολα της Ευρώπης. Πόσο πολύπλοκες είναι οι πολιτικές λύσεις, πόσο κοπιαστική η διαδικασία, νομίζω αυτό το ξέρετε εσείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλύτερα από όλους. Εδώ πέρα συναντιούνται αντικρουόμενα συμφέροντα, αλλά και διαφορετικοί πολιτισμοί, γλώσσες και παραδόσεις. Η ποικιλομορφία της Ευρώπης είναι μια περιπέτεια, αλλά είναι και κουραστική. Και θεωρώ πως ε, συμφωνούν εδώ πέρα και ο Αντώνιο και οι επικεφαλής των ε, ομάδων. Αλλά γι' αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε περισσότερο σήμερα την Ευρώπη. Δεν πρέπει ο καθένας να περιχαρακωθεί με τους ομοειδεάτες του. Πρέπει να ξεπεράσουμε το μικρό περιβάλλον μας ο καθένας. Δεν επιτρέπεται να ξαναγυρίσουμε στην εθνική μας γωνιά. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε ακριβώς να ξεπεράσουμε αυτά τα οποία μας χωρίζουν. Και βεβαίως αυτό σημαίνει και σήμαινε πάντα η, σημαίνει ότι και οι άλλοι μπορεί να έχουν δίκιο η Ευρώπη ιδρύθηκε με βάση την υπόθεση ότι και ο άλλος μπορεί να έχει δίκιο. Η Ευρώπη πάντα πετύχαινε συμβιβασμούς. Οι επιτυχίες της Ευρώπης ήταν πάντα οι δύσκολες αλλά ειρηνικές εξισορροπήσεις των συμφερόντων. Αυτό συμβολίζει αυτό το κοινοβούλιο, τα 28 έθνη. Ποιος θα γίνει βουλευτής χωρίς να έχει την θέληση να πείσει αλλά ταυτόχρονα και την θέληση να πιστεί. Χωρίς να έχει πάθος για το δύσκολο, για τον κόπο της δημοκρατίας. Όλοι σε αυτή την αίθουσα έχετε τον μεγάλο σεβασμό μου και την στήριξή μου κύριε και κύριοι. Την στήριξή μου γιατί γνωρίζω πως υπάρχουν και αρκετές άλλες δυνάμεις οι οποίες είναι έτοιμες πάντα με απλές απαντήσεις που θεωρούν ότι θα πρέπει να υπάρχει το ισχυρό χέρι. Βλέπουμε ξανά να αυξάνεται η γοητεία του αυταρχισμού όχι μόνο για τη δυτικά και ανατολικά των ευρωπαϊκών συνόρων σημαίνει αυτό, αλλά και εδώ, στη μέση της Ευρώπης. Οι λαϊκιστές οι οποίοι παρουσιάζουν τον κόσμο άσπρο-μαύρο και κεφαλαιοποιούν τον φόβο. Βεβαίως, προσπαθώ πάντα να μην κινδυνόλογο. Το κοινοβούλιο αυτό μπορεί να αντέξει τις διαφωνίες και τις χρειάζεται, αλλά όποιος απορρίπτει τα κοινοβούλια και την δημοκρατία ως σπατάλη χρόνου, όποιος θεωρεί ότι ο συμβιβασμός είναι αδυναμία και όποιος δεν ξεχωρίζει τα γεγονότα από το ψέμα, κλονίζει τα θεμέλια της δημοκρατίας και θα πρέπει να μας βρει απέναντι. Ο κόσμος στον οποίο ζούμε έχει γίνει λιγότερο ασφαλής και πιο περίπλοκος. Πολλοί κόσμος ανησυχεί για το μέλλον. Φοβάται ότι χάνει τον έλεγχο. Και βεβαίως κλείνει έτσι πιο εύκολα στις φωνές εκείνες που του λένε έλα πίσω, πίσω από τα τείχη του έθνους. Να κλείσουμε τα σύνορα, μόνο έτσι θα ξανακερδίσουμε την κυριαρχία μας. Αλλά δεν είναι μόνο άφελες, είναι ανέθινο να λέμε στον κόσμο ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κινδύνους όπως τρομοκρατία ή κλιματική αλλαγή με τείχη και μπάρες. Είναι ανεύθυνο να παριστάνουμε ότι σε έναν κόσμο που γίνεται όλο πιο περίπλοκος οι απαντήσεις γίνονται απλούστερες. Και είναι λάθος να λέμε ότι σε αυτό τον κόσμο μπορεί με ευρωπαϊκή χώρα μόνη της χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση να ακουστεί ή να επιβάλλει τα οικονομικά της συμφέροντα. Αντιθέτως, κυρίες και κύριοι, αν η Ευρώπη δεν γίνει παγκόσμιος παίχτης, τότε θα γίνουμε όλοι παιχνίδι στα χέρια άλλων δυνάμεων. Και μάλιστα αυτό εννοούσε πιθανότατα ο Μάικλ Χέζελτάιν, ειδικά ένας Βρετανός, όταν είπε ότι το Brexit είναι η μεγαλύτερη απώλεια κυριαρχία της Βρετανίας που είχε ζήσει. Και έχει δίκιο. take back control, να πάρουμε τον έλεγχο. Είναι πράγματι ισχυρό σύνθημα, αλλά να σας πω, οι εθνικιστές δεν θα το τηρήσουν. Αν μπορεί να τηρηθεί, μπορούμε να το τηρήσουμε εμείς από κοινού. Αν δεν επιρρύπτουμε όλες τις ευθύνες στις Βρυξέλλες, αλλά τις ασκούμε από κοινού. Αν ενισχύσουμε την εσωτερική αγορά και ταυτόχρονα προστατεύσουμε αυτούς οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έζησαν την αρνητική πλευρά της παγκοσμιοποίησης ιδιαίτερα. Αν ενισχύσουμε την καινοτομία και τη δημιουργικότητά μας έτσι ώστε η Ευρώπη να διαμορφώσει την αλλαγή και να μην την υφίσταται μόνο. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να νικήσουμε τους λαϊκιστές και να πούμε ότι δεν χάνουμε κυριαρχία στην Ευρώπη. Το αντίθετο. Κερδίζουμε κυριαρχία και δύναμη και ειδικό βάρος στον κόσμο. Η κρίση, κυρίε και κύριοι, είναι μια ευκαιρία να δούμε την Ευρώπη όπως είναι. Πραγματικά, χωρίς ψευδεστήσεις, χωρίς υπερβολική αισιοδοξία, με όλα τα ισχυρά και ανίσχυρα σημεία της. Και μας αναγκάζει να απαντήσουμε στο ερώτημα ποια και πόση ευρωπαϊκή ενοποίηση θέλουμε. Λευκή Βίβλος της Κομισιόν μας προσφέρει κάποιες επιλογές. Βεβαίως ένα νομίζω είναι σαφές, ότι το μόνιμο αυτομπλοκάρισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η χειρότερη δυνατή επιλογή. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε από κοινού, δεν μπορεί τελικά ο καθένας να κερδίσει 100%. Είναι πολύ πολύπλοκα τα προβλήματα και οι προσδοκίες μας είναι πολύ διαφορετικές. Ναι, Θέλουμε μια ισχυρότερη Ευρώπη και περισσότερες ευρωπαϊκές λύσεις, αλλά πρέπει να αφήσουμε και περιθώριο για εκείνα τα κράτη-μέλη τα οποία δεν θέλουν να ακολουθήσουν ή δεν μπορούν να ακολουθήσουν κάποια βήματα ενοποίησης. Ναι, να είμαστε αλληλέγγυοι με χώρες οι οποίες υποφέρουν από την οικονομική κρίση και πρέπει να κάνουν σκληρές μεταρρυθμίσεις, αλλά η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη μπορεί να συμπληρώσει μόνο, δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις εθνικές προσπάθειες. Ναι, να βοηθήσουμε ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν από πόλεμο και διώξεις, αλλά επειδή και οι κοινέ μας δυνατότητες είναι πεπερασμένες, πρέπει να αποφασίσουμε πόση ευθύνη θα φέρει ο καθένας. Ναι, θέλουμε να υπάρχει εσωτερική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά γνωρίζουμε η Ευρώπη είναι μεγαλύτερη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν δεν είμαστε σε επαφή και με τους γείτονές μας ε, προς Ανατολάς και προς Νότον δεν θα έχουμε ποτέ ειρήνη σε αυτή την Ήπειρο. Ναι, κυρίες και κύριοι, κανένα από αυτά τα προβλήματα δεν είναι απλό. Και δεν μπορούμε να αγνοούμε τους φόβους των ανθρώπων, αλλά αυτοί οι οποίοι οικοδόμησαν την Ευρώπη είχαν να αντιμετωπίσουν πολύ πιο δύσκολα προβλήματα και αντικατέστησαν το πεδίο της μάχης με την Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων και την αντιπαράθεση μέσω της ειρηνικής εξισορρόψης των συμφερόντων. Αποδείχθηκαν έξυπνοι και λογικοί και ο σημερινός κόσμος, ένας κόσμος γεμάτος αβεβαιότητα, δεν μας επιτρέπει να είμαστε λιγότερο έξυπνοι από ότι οι προκάτοχοί μας. Δεν είναι το πρόβλημα, το ποια είναι τα προβλήματα που πρέπει να λυθούν. Αυτό είναι σαφές. Αυτό το οποίο λείπει είναι το θάρρος και η βούληση να λυθούν στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Βεβαίω, όταν μιλάμε για εξορρόπηση συμφερόντων, υπάρχει και διαφωνία. Διαφωνούμε στην Ευρώπη και αυτό δεν είναι σημάδι ε, παρακμής. Και εγώ βεβαίως τα τελευταία 25 χρόνια α, της ε, πολιτικής είμαι μαθημένος σε αυτά. Αλλά όταν τσακωνόμαστε και διαφωνούμε στην Ευρώπη το κάνουμε με βάση κάποια θεμέλια. Πάρα πολλά θέματα είναι περίπλοκα αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε τα στοιχειώδη, τα σημαντικά, η ελευθερία και η δημοκρατία το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι προς διαπραγμάτευση. Αυτό αναφέρεται και στο άρθρο 2 της συνθήκης της Ένωσης και δεσμεύει όλα τα κράτη-μέλη. Αυτός είναι ο πυρήνας της Ευρώπης. Αυτό ακριβώς αντιπροσωπεύει η Ευρώπη στα μάτια του κόσμου και αυτό ζηλεύουν πολύ. Αν λοιπόν επιμένουμε σε αυτό, αν θέλουμε να είμαστε ένας φάρος κράτους δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο. Τότε δεν μπορούμε να αδιαφορούμε όταν πραγματικά αυτά τα θεμέλια τρίζουν. Και βλέπουμε και δεν μπορούμε να είμαστε αδιάφοροι όταν βλέπουμε ότι η κοινωνία των πολιτών ή ακόμα και η επιστήμη καταπιέζεται όπως γίνεται τώρα στο Κέντρο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Βουδαπέστης. αλλά βεβαίως ο επίμαχος είναι και ο ρόλος της δικής μου χώρας. Κάποιοι ζητούν από τη Γερμανία να παίξει πιο ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη, άλλοι προειδοποιούν για γερμανική κυριαρχία. Και ο νέο εκλεγής πρόεδρος του σημαντικότερου συμμάχου μας είπε προσφάτως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι παρά ένα όχημα κυριαρχίας Γερμανίας. Πρόκειται για παρεξήγηση. η δύναμη της Ευρώπης δεν μπορεί να υπάρξει υπό την ηγεσία ενός, αλλά υπό την ευθύνη όλων. Και βεβαίως η Γερμανία ως μεγαλύτερη και πολυπληθέστερη χώρα έχει μια ιδιαίτερη ευθύνη. Αλλά γνωρίζουμε τα όρια των δυνατοτήτων μας. Και δεν θα ξεχάσουμε πως και οι άλλοι, όπως είπα, μπορεί να έχουν δίκαιο στην Ευρώπη. Γνωρίζουμε τι οφείλουμε στην Ευρώπη και η Ενωμένη Ευρώπη είναι η επιτυχημένη απάντηση στην ιστορία μας και την γεωγραφία μας. Για μας τους ίδιους και για τους γειτονές μας. Και νιώθουμε ότι μια ισχυρή Ευρώπη δεν είναι μόνο προς το κοινό μας συμφέρον, αλλά ότι είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας πλέον. Γι' αυτό πρέπει να ξέρετε το εξή. Οι Γερμανοί θέλουν να διατηρήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλουμε να έχουμε ένα κοινό μέλλον στην Ευρώπη και αποκοινούμε τους εταίρους μας μεγάλους και μικρούς να προχωρήσουμε ισότιμα και με τις ίδιες υποχρεώσεις. Αλλά πέρα από κάθε εθνικό συμφέρον υπάρχει κάτι το τελείως διαφορετικό και πολύ σημαντικότερο. Όχι για όλους, αλλά για τους περισσότερους ανθρώπους στην Γερμανία η Ευρώπη είναι κάτι το οποίο αγαπούν. Γι' αυτό σας διηγήθηκα και την προσωπική μου ιστορία σε σχέση με την Ευρώπη. Γι' αυτό ακριβώς και τις ε, τελευταίες εβδομάδες πολλοί νέοι στην Ευρώπη διηγήθηκαν την ιστορία της δικής τους Ευρώπης. Και οι νέοι είπαν ότι βαρέθηκαν να μιλούν για την Ευρώπη μόνο όσοι την κακολογούν. Δεν θέλουν το μέλλον τους να το κλέψουν οι λαϊκιστές ή να καταστραφεί λόγω αδράνειας. Γι' αυτό ακριβώς είδαμε ότι ο σφιγμός Ευρώπης χτυπάει στους δρόμους και στις πλατείες. και ακόμα και αν η δικιά μας γενιά δεν το λέει έτσι. Για πολλά από τα παιδιά και τα εγγόνια μας η Ευρώπη πλέον είναι μια δεύτερη πατρίδα. Οι νέοι αυτοί γνωρίζουν πως δεν είναι αντίφαση το να τη χώρα τους και ταυτόχρονα να είναι Ευρωπαίοι. Και έχουν δίκιο οι νέοι. Τέλος, πέρσι έκανα ένα ιδιωτικό ταξίδι με την οικογένειά μου στον Πρέσλα ήθελα να δω την πόλη που γεννήθηκε η μητέρα μου. Γιατί τη γνώριζα μόνο από τις άσχημες αναμνήσεις της. Μου είχε διηγηθεί τις ιστορίες του πολέμου και της φυγής στην Δύση με μητέρα, θεία, αδερφή και 7 παιδιά. Ο εθνικισμός και οι συνέπειές του σημάδεψαν τη ζωή της μητέρας μου και με αυτόν τον τρόπο σημάδεψαν και την εικόνα που είχα εγώ για την πόλη της. Και όμως πέρσι, το 2016, πήγαμε σε μια τελείως διαφορετική πόλη. Μια πόλη που ήταν πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης και έλαμπε με συζητήσεις, με μουσική στους δρόμους, στις πλατείες όπου νέοι από το Βίλνιου, στο Βούπερταλ και την Βερόνα γιόρταζαν την Ευρώπη. Κυρίε και κύριοι, εκεί πέρα δεν υπήρχε καθόλου στενομιέλια. Εκεί ζούσε το όνειρο του ευρωπαϊκού μέλλοντος. Και τώρα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, επαφείτε σε εμάς να μην σταματήσει το ευρωπαϊκό όνειρο. Αυτό είναι το μήνυμα που σας φέρνω από τη χώρα μου. Ναι, θέλουμε την Ευρώπη, θέλουμε να οικοδομήσουμε μια καλύτερη Ευρώπη και θέλουμε να είμαστε μια ευρωπαϊκή Γερμανία. Σας ευχαριστώ. Να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας που απεδέχθη την πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έκανε μια παρουσίαση η οποία θα λειτουργήσει σαν κίνητρο για τις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν και όλες τις επόμενες εβδομάδες η Ευρώπη θα πρέπει να αλλάξει, θα πρέπει να διορθωθεί. Νομίζω ότι αυτό είναι το θετικό μήνυμα το οποίο απέστειλε ο πρόεδρος Στάινμαγερ. Και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το μήνυμα αυτό.